Morning, dear Καλημέρα συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Περνάμε στο σημείο 6 της ημερησία ε, διάταξη προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και καταπολέμηση τη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Εισηγητή ο Βέρνερ Λάγκεν θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Σα δίνω λοιπόν αμέσω τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεσης ε, ασχολείται κυρίως με την ε, έκθεση της ε, Κομισιόν για τις 7 Απριλίου για το πολιτές σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα της απάτης ΦΠΑ. Ο κύριος Μοσκοβισή υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης το οποίο πηγαίνει προς μια σωστή κατεύθυνση αλλά βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα κύρια προβλήματα. Δηλαδή την τεράστια απάτη που φτάνει σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος. Μιλάμε για μια σημαντική πηγή εσόδων, 7% του ε, ΑΕΠ, ένα 3 εκατομμύριο ευρώ και με 17% ποσοστό απάτης ε, έχουμε ένα ποσοστό το οποίο δεν ε, μειώνεται και αφορά και και απάτη αλλά και εντός των κρατών μελών και το παλεύουμε εδώ και χρόνια χωρίς μεγάλα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν τώρα το σχέδιο έκθεσης που υπάρχει σε όλες ε, τις γλώσσες έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα τα σημαντικότερα πράγματα. Από το 1993 στις σχετικές διατάξεις οδηγίας αναφέρεται πως θα πρέπει να υπάρξει ένα οριστικό καθεστώς, γιατί μέχρι τώρα ήταν μεταβατικό. Έχουν περάσει λοιπόν 23 χρόνια, οπότε ο κύριος ε, Μοσκοβισή θέλει μετά από 25 χρόνια το 2018 να έχουμε επιτέλους ένα οριστικό σύστημα. Το οριστικό σύστημα θα πρέπει να έχει στόχο τα αποτελέσματα. Το τωρινό σύστημα λόγω των πολλών απατών έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Υπάρχει ήδη μια γνωμοσύνη η οποία αναπτύσσει πέντε εναλλακτικέ και μας λέει ποιες θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν την γραφειοκρατία και την απάτη. Και ο κύριος ε, Μοσκοβισή από αυτές τις πέντε εναλλακτικέ, μας υπέβαλε δύο μόνο για συζήτηση, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε. Διαπιστώνουμε πως η συνεργασία των κρατών μελών δεν ήταν καλή στο παρελθόν δεν υπήρχαν επαρκείς ανταλλαγές ε, στοιχείων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν εύκολη απάτη καρουζέλ, η λεγόμενη, δηλαδή κάποιος ε, βλέπε, εισπράττει το ΦΠΑ στη μια χώρα και δεν φαίνεται πουθενά αυτό στην άλλη χώρα και από αυτό μιλάμε τουλάχιστον για 50 δισεκατομμύρια και βλέπουμε πως ε, τα κράτη-μέλη εδώ πέρα δεν έχουν κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε. Γι' αυτό Σωστά προτείνει ο κύριος Μοσκοβισή να χρησιμοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία έτσι ώστε οι πληροφορίες να μεταδίδονται ταυτόχρονα από το ένα κράτος στο άλλο και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες επιτρέπουν ε, ξαφνικά να πληρώνει τον ΦΠΑ ο τελικός ε, καταναλωτής και αυτός μετά να εξαφανίζεται. Επίσης, αναφέρεται πως ε, το οριστικό σύστημα θα πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες για το τι γίνεται στην χώρα ε, προέλευσης. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το τι γίνεται στην χώρα προορισμού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ανεξαρτήτως του τι, από πού προέρχεται το αγαθό, επιβάλλεται ο ΦΠΑ της χώρας ε, προορισμού. Αυτό είναι ένα σύστημα ουδέτερο προς τον ανταγωνισμό, ενώ η αρχική πρόθεση για την ε, χώρα προέλευσης είχε νόημα μόνο αν δεν υπάρχει μεγάλη ψαλίδα στο ΦΠΑ μεταξύ των χωρών. Θυμάμαι πριν από 15 χρόνια ήδη υπήρχε αυτή η συζήτηση και εκεί πέρα η Κομισιόν πρότεινε να υπάρχει μια ψαλίδα το πολύ 4% μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου ΦΠΑ για να μην υπάρχει στρέβλος του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει όμως πλειοψηφία για την χώρα, της, ε, για τη χώρα προέλευσης στο Συμβούλιο, οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός για την χώρα προορισμού. Μετά υπάρχει το επόμενο θέμα που είναι τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ, τα οποία είναι εν μέρη παραδοσιακά. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουμε και μηδέν. Μπορείτε λοιπόν, έχω εδώ πέρα τον κατάλογο και να ρωτιέται κανείς γιατί τα κτηνιατρικά φάρμακα από το στόμα στην Ιρλανδία φορολογούνται με μηδέν ή πωλήσει διαφόρων οργανώσεων στη Φιλανδία ή παραδείγματο χάρη δανεισμός ε, άτοκος ε, σε ενώσεις ε, τυφλών. Ένας πάρα πολύ εκτεταμένος κατάλογος αλλά θα πρέπει τελικά τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο, όχι σε κοινό ποσοστό ΦΠΑ. Να δουν δηλαδή ποιε ε, υπηρεσίες ε, θα έχουν χαμηλό ΦΠΑ ή θα απαλλάσσονται κιόλας. Αυτό το είδε λοιπόν το δικαστήριο και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αποτελούν μέσω κοινωνικής πολιτικής, αλλά ότι επιτρέπονται για τα τρόφιμα. Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να επανεξεταστεί. Μετά. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Το θέμα του πώς ε, θα γίνεται η ε, παράδοση, αν θα γίνεται ψηφιακά ή φυσικά. Και εκεί πέρα υπάρχει μια απόφαση για, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν έχει καμία σημασία. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ο ίδιος. Γνωρίζουμε τι γίνεται με το Amazon στο Λουξεμβούργο. Οπότε θα πρέπει εδώ πέρα οπωσδήποτε να υπάρξει το ίδιο ύψος ε, ΦΠΑ. Το επόμενο θέμα βεβαίως είναι η πρόταση να υπάρξει μια αντίστροφη χρέωση, κατά το οποίο σημαίνει πως όπως τώρα θα πληρώνει ο ΦΠΑ το, συνολικό, το, το τελικός πελάτης στο συνολικό ποσοστό ΦΠΑ, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει πως ε, όταν υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουμε προβλήματα φορολογικά, εφοδιαστικά κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθούν αυτά τα βήματα και ειδικά στις διασυνοριακές συναλλαγές να υπάρξει καλύτερο συντονισμός των αρμοδίων αρχών και αυτό το σύστημα της αντίστροφης χρέωσης ήδη υπάρχει σε κάποιους ε, κλάδους εκεί δηλαδή όπου έχουμε υψηλό ποσοστό απάτης εκεί έχει εισαχθεί αυτό το σύστημα και υπάρχει ένα αίτημα της τσεχικής κυβέρνησης ε, το οποίο εξετάζει η Ολλανδική Προεδρία και το στηρίζει το τελευταίο εξάμεινο σύμφωνα δε με το οποίο σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν υπήρξε μια θετική αξιολόγηση. Γι' αυτό προτείνω να γίνει μια επιστημονική μελέτη και να το δούμε σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις ε, για την χώρα προορισμού. Το τελευταίο το ανέφερα αφορά την γραφειοκρατία που είναι πάρα πολύ επιβαρυντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι τόσο εύκολο του να κάνουν διάκριση μεταξύ των παραδόσεών τους ανάλογα με το κράτος μέλος αλλά την άλλη πρέπει να πληρώσουν τον φόρο τη μέρα την οποία πρέπει να τον πληρώσουν αλλά μετά η επιστροφή του ΦΠΑ είναι ένα άλλο ζήτημα και τα κράτη προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες. Οπότε το σύστημα αυτό της αντίστροφης χρέωσης ε, θα τα απλοποιήσει όλα αυτά. Τελευταίο. Εγώ θεωρώ πως υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ε, απολύτως αναγκαία. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα εδώ και στα βασικά αυτά ζητήματα θα πρέπει να ακολουθηθεί η τακτική νομοθετική διαδικασία και δεν απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ξέρω βεβαίως πως αυτό σημαίνει αλλαγή της συνθήκης, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι μας εμποδίζει να καταπολεμήσουμε την απάτη του ΦΠΑ. Τελευταία λέξη. Εγώ δεν θέλω να καθορίσω ανώτατα ή κατώτατα ποσοστά και να μπω στα χωράφια των κρατών μελών. Αλλά χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση, σύγχρονες ε, μέθοδοι και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί αυτοί οι οποίοι κλέβουν ε, τον ΦΠΑ είναι τόσο επιδέξοι και ποιο είναι το αποτέλεσμα οι νόμιμοι οι οποίοι δεν μπορούν να τον αποφύγουν φέρουν το βάρος των υπολείπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η Ελίζα Φερέιρα τώρα έχει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλάω εκ μέρους του κύριου Ζάνε, του σκιώδου εισηγητή που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, επειδή έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις εκτός Βρυξελών. Μου ζήτησε λοιπόν να μιλήσω εδώ εκ μέρους του. Κάτι το οποίο κάνω με χαρά. Το θέμα αυτό πιστεύω ότι είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό και χαίρομαι για την έκθεση αυτή που εξετάζουμε σήμερα που μας παρουσίασε ο κύριος Βέρνερ. Η έκθεση ανταποκρίνεται σε ένα στόχο κλειδί που είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστούν ώστε σταματήσει πια ένα σύστημα το οποίο σήμερα είναι απλώς απαράδεκτο. Ένα σύστημα δηλαδή διευρυμένης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Ο στόχος κλειδί λοιπόν, αυτό που πρέπει να πετύχουμε, αυτό που πρέπει να φτιάξουμε μαζί, είναι μια ισχυρή θέση έτσι ώστε να σταματήσει ένα καθεστώς συναλλαγών που ισχύει εδώ και 23 χρόνια. Χρειάζεται μια πλήρης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ΦΠΑ. Έτσι θα σταματήσει αυτό το σκάνδαλο της απάτης του ΦΠΑ και της έμεσης φορολόγησης γενικότερα. Συνεπώς, από κοινού, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να δουλέψει σκληρά. Έχουμε δει διάφορες μελέτες να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια που προτείνουν λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενστενιστεί κάποιες από αυτές τις ιδέες και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι Έχουμε φτάσει όμως στο σημείο που πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, τις αποχρώσεις, γιατί μερικές φορές είναι σημαντικές. Οι αλλαγές λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Φυσικά και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά και συμφωνώ με τον εισηγητή για το ότι πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί συγχρόνως. Δεν πρέπει να βάλουμε τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να συζητήσουμε κατάλληλα όλες τις λεπτομέρειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα θέματα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Όσον αφορά το εύρος των προϊόντων που καλύπτονται από μειωμένο ΦΠΑ, εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές και πρέπει να τις επεξεργαστούμε όλες προσεκτικά. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε βασικά προϊόντα, τα οποία σήμερα καλύπτονται στο οποίο επιβάλλονται πολύ υψηλές τιμές ΦΠΑ σε ορισμένες χώρες και σε άλλες έως και καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν όλες τις επιλογές πρέπει να τις κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά. Το θέμα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού. Όμως δεν θα πρέπει όλες τις προσπάθειές μας να τις βάλουμε σε αυτό το καλάθι, δεν πρέπει να χάσουμε υπερβολικό χρόνο πάνω σε αυτό, ενώ πρέπει από την άλλη να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροπάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροποφυγής. Τονίζω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα αποτελεί ένα εμπόδιο στην πρόοδο που θέλουμε να επιτευχθεί και όσον αφορά την άμεση και όσον αφορά την έμεση φορολογία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε την κατάσταση δεδομένη της πρόοδου που έχει επιτευχθεί με την ενιαγορά και το ενιονόμισμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλα αυτά πώς αναφέρονται και στη συνθήκη, γιατί η ομοφωνία στο Σεβούλιο δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση για τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαλούκα από το ECR τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να δράσουμε γρήγορα γιατί το ύψος της απάτης είναι τεράστιο. Δεν ξέρω πού βρήκατε αυτά τα νούμερα αλλά η τάξη του μεγέθους είναι πολύ ανισχυτική. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποια δισεκατομμύρια πάνω κάτω για το μέγεθος, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, σημαίνουν τα νούμερα αυτά ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Γι' αυτό χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν ε, υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερε ο προλαλής ε, τα 23 χρόνια δηλαδή. Χαιρετίζω επίσης το ότι η Κομισιόν ε, επιτέλους αποφάσισε οριστικά να οριστεί η χώρα προορισμού ως βάση υπολογισμού κατά το οποίο είναι ουδέτερο ως προς τον ανταγωνισμό για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα κατά το οποίο δεν θα ήταν ένα σύστημα με την ε, χώρα προέλευσης. Γι' αυτό απορώ που άργησε τόσο πολύ η Κομισιόν επίσης στηρίζουμε ρητός ε, το ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εφαρμόσει την αρχή αυτή τώρα σύνεπως. Μετά ο κύριος Λάγγεν είπε ότι υπάρχουν επιστημονικές έρευνες ε, που αναφέρουν διάφορες δυνατότητες διαμόρφωσης του συστήματος του ΦΠΑ και η Κομισιόν επέλεξε να αγνοήσει κάποιες από αυτές και να ακολουθήσει κάποιες άλλες. Θετικό το ότι ο κύριος Λάγγεν μας λέει πως είναι προβληματική η κατεύθυνση που παίρνει η Κομισιόν και ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις ε, όσον αφορά, η διαδικα... όσον αφορά την συλλογή του ΦΠΑ, παραδείγματο χάρη η διαδικασία της αντίστροφης χρέωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είστε ακόμη πιο θαραλέως όχι μόνο να ζητήσουμε εξέταση των ε, άλλων ε, πρακτικών, οι οποίες είναι δοκιμασμένες και στην πράξη, αλλά πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα και να πούμε πώς θα πρέπει να ακολουθηθεί και να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία της αντίστροφης χρέωσης. Θα ήθελα να πω πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των αποφάσεων επί της αρχής ε, της ε, κατεύθυνσης που θα πάρει το σύστημα, δηλαδή η χώρα προέλευσης ή χώρα προορισμού και πρέπει πράγματι να είμαστε υπέρ της χώρας προορισμού και να το χωρίσουμε μετά από το πώς θα γίνεται η συλλογή του ΦΠΑ, γιατί ε, το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της μίας ή της άλλης χώρας και να έχουμε παραδοσιακή αντίστροφη χρέωση. Δεν υπάρχει επίσης ε, κανένα πρόβλημα να επιλέξουν ελεύθερα τα κράτη-μέλη ποια διαδικασία θέλουν. Οπότε, μια που απαιτείται και ομοφωνία για να αλλάξει σχετική οδηγία, εγώ ζητάω να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία. Και το θέμα του πώς θα συλλεγεί ο ΦΠΑ θα πρέπει να αφαιθεί. Και κάποια κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν την παραδοσιακή, κάποια άλλη την αντίστροφη χρέωση, ανάλογα με το πόση εμπιστοσύνη έχουν στις διάφορες φάσεις ε, της εμπορικής αλυσίδας και πόσο υψηλή εκτιμούν ότι είναι η πιθανότητα απάτης από ό,τι σε σχέση με την τωρινή διαδικασία. Οπότε νομίζω πως ε, μπορούμε να αφήσουμε αυτή την απόφαση στα κράτη-μέλη. Οπότε αυτό το οποίο θα ζητούσα εγώ είναι να ξέρουμε πως η νομοθετική πρόταση πρέπει να πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να απαριθμούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για να υπάρχει ευελιξία, όπως είπαμε, στο επίπεδο των κρατών μελών. Όσον αφορά τώρα του, τον μειωμένο ΦΠΑ, θα πρέπει τα κρατημέλη να είναι ελεύθερα να καθορίζουν ε, το ύψος του ΦΠΑ, αλλά βεβαίως για λόγους διαφάνειας καλό θα ήταν να γνωρίζουμε και να μειωθεί ο αριθμός των ε, προϊόντων και υπηρεσιών που ε, υπάρχουν σε μειωμένο ΦΠΑ. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να αλλάξει η συνθήκη, ούτε να φύγουμε από την ομοφωνία σε θέματα φορολογίας. Είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τελειώνω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα, με αυτό το σημείο της έκθεσης δεν μπορώ να συμφωνήσω και δεν χρειαζόμαστε αλλαγή της συνθήκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεζακ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ αξιολογή η εκθέση που έχουμε ενώπιόν μα και ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους και η συζήτηση έχει προχωρήσει σε βάθος και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα περισσότερα σίγουρα. Ε, ε, το μέγεθο της απάτης έχει διαστάσεις σκανδαλώδε και ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Και ακριβώ όπω είπε και ο εισηγητής, Έχουμε αυτή την προσπάθεια της ε, Προεδρίας για τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης και αυτό είναι το, το μόνο που έχουμε προς το παρόν, το μόνο που πρόσφατα έχει προκύψει. Άρα δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο τις ε, σχετικές μελέτες, αλλά όπως λέγεται το σχέδιο κειμένων, θα πρέπει να γίνονται κάποιες ε, προσπάθειες για κάποια πιλωτικά προγράμματα, όπως έγινε και στο Συμβούλιο, για αυτή τη διαδικασία της αντιστροφής της χρέωσης. Ε, επίσης, νομίζω ότι με αυτή την προσέγγιση θα εξαλαφρώσουμε και θα ανακουφίσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ε, βάρος της γραφειοκρατίας. Άρα χρειάζεται και συνεργασία των μελών και γενικότερα για όλη αυτή την προσέγγιση και για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερη ελευθερία τα κράτη-μέλη για να έχουν κάποιον μειωμένο συντελεστή. Αυτό είναι καλή ιδέα. Και γενικώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σωστή κατεύθυνση και πάλι ευχαριστίες προς όλους τους αδέλφους και τον γιατί, ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για την ε, Γκουέ, κυρία Μπερμέχο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το σημερινό σύστημα είναι άτυπο και είναι αποτελεσματικό. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Και συμφωνούμε με τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για μας το πρόβλημα δεν είναι απλώς διοικητικό, είναι πολιτικό. Άρα χρειάζεται να προβληματιστούμε για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο φόρος και να δούμε τι θα γίνει με τις κοινωνικές επιπτώσεις. Ο μειωμένος συντελεστής για βασικά προϊόντα, γιατί πρώτες ανάγκες για κάποια ε, προϊόντα κοινή χρήση και κάποια πολιτιστικά θα πρέπει ε, εκεί οι φτωχότεροι να δίνουν λιγότερα. Και γιατί πρόκειται για την προσβασιμότητα σε κάποια αγαθά πάρα πολύ σημαντικά. Ε, άρα θα πρέπει να φορολογηθούν οι πλουσιότεροι και τα είδη πολυτελείας να έχουν αυξημένο συντελεστή. Ε, ε, ε, Όπω διφόρμα τα λέει η Κομισιόν, δεν θα πρέπει να παρατηρούμε το σημερινό καθεστώ. Θα πρέπει να είναι προοδευτικό αυτό ο φόρο. Δεν θα πρέπει να, να είναι βασιλιά ο, ο ανταγωνισμός και η διακυβέρνηση αγοράς. Δεν θα πρέπει να αυξάνουμε την ανισότητα μεταξύ των φορολογουμένων. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε προοδευτικό φόρο και έχουμε και απάτη από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν θα τα προβλήματα τα οποία τα ε, επισημάνει η Κομισιόν σαν και ένα στο νόμο πρώτα πρώτα. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε και έτσι να αντιμετωπίσουμε οριστικά την απάτη και άλλα μέτρα είναι αναγκαία ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διοίκηση, οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους και έτσι θα πολεμήσουμε την απάτη και θα πρέπει η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρα σε αυτό το μέτωπο γιατί όταν έχουμε επιθεωρήσεις απονευρωμένες όταν δεν διατίθενται οι απαραίτητοι Πόρει αυτό δεν μας οδηγεί σε φορολογική δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό γίνεται και στη χώρα μου. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τώρα για τους ε, πρασίνους. Έχετε το λόγο. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικά διάφορα που θα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμεριζόμαι αυτό που λέει για κατηγορίε τη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Επιτροπή ότι θα πρέπει το διοικητικό κόστο να μην μειωθεί όσον αφορά τι ΜΜΕ. Και σήμερα βλέπουμε υπάρχει μια πολυνομία, πολύπλοκα συστήματα, πολλέ παρεκκλήσει να αφορμούν του συντελεστέ. Και για αυτό είμαστε υπέρ του να έχουμε ενιαίο σύστημα επί τη βάση της αρχής του προορισμού. Και θεωρούμε ότι έχει τη σωστή ερώτα η πρόταση της Κομισιόν, αλλά βέβαια όλα τα υπέρ και τα κατά θα πρέπει να τα ζυγίσουμε. Αυτή η μόνο απευθυντική θηρίδα για το νέο σύστημα θα πρέπει να ενισχυθεί με τα συμπράσματα που έχουμε από το ίδιο σύστημα που έχουμε για τα ψηφιακά. Ε, Αλλιώ θα στριμωχτούν οι επιχειρήσει και στη χώρα μου και Οπότε θα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι ε, μικρέ ε, επιχειρήσει οι οποίε θα αναγκαστούν είτε να σταματήσουν το εμπόριο ή να κλείσουν. Γιατί αυτό συνέβη και στη δική μου περιφέρεια. Για τις ΜΜΕ χρειάζεται κάποιο είδους αντιστάθμιση, κάποιο είδους αρρωγή για να προσαρμοστούν στο καινούργιο σύστημα θα πρέπει οι ΜΜΕ να εμπλακούν στην προετοιμασία αυτού του πακέτου ΦΠΑ. Οι μειωμένε συντελεστέ για διάφορα αγαθά είναι θέμα δύσκολο. Το είπαν και οι προλαλήσαντε. Έχει δύο επιλογέ εδώ. Η Κομισιόν μα λέει ή θα πρέπει να αναθεωρήσει τον σημερινό κατάλογο των προϊόντων ή να δώσει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να επιλέξουν πού θα εφαρμόσουν τον μειωμένο συντελεστή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν και τα υπέρ έχουμε λιγότερες εξαιρέσεις, περισσότερη εναρμόνιση, αλλά από την άλλη μεριά είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν κάποια διακριτική ευχαίρεια να διαλέξουν τους μειωμένους συντελεστές ανάλογα με τις παραδόσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις και σύμφωνα με την αρχή της επιφύλαξης. Ε, Βεβαίω, α όχι λάθος, λάθος, δεν είναι για την... Ε, δεν η επιφύλαξη, είναι η επικουρικότητα που μετράει εδώ. Άρα χρειάζεται τέτοια προσέγγιση ε, για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους βιωσιμότητας ε, σε αυτά τα προϊόντα ε, ε, όπως και για τα ταμπών για τις κυρίες αυτά θα πρέπει να έχουν μειωμένο συντελεστή και άρα θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία, άρα θα πρέπει να σχεδιαστεί το σύστημα έτσι, ούτω ώστε να μην έχουμε προσφυγή στα δικαστήρια, να μην υπάρχει ανταγωνισμός φορολογικός. Έτσι θα αποφύγουμε τους κινδύνους και θα πρέπει επομένως να τα βρουν οι χώρες στο Συμβούλιο. Χρειάζεται επομένως πανευρωπαϊκή ε, πολιτική, χρειάζεται συντονισμός και τελικά να καταλήξουμε σε τέτοια αποτέλεσμα που θα βοηθήσουν την υγεία, το περιβάλλον και να μην ε, υπάρχει κατανάλωση περισσότερη βλαπτικών προϊόντων. Ε, έχουμε δεδομένες τις μελέτες που ξεκίνησαν το 2008 και έχουμε τώρα στο Συμβούλιο πραγματεύσεις, άρα θα πρέπει όλες αυτές οι πολιτικές να ξαναμπούν στο θεματολόγιο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάνη ήρθε, όχι. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Τότε πάμε στο Κάτσο Διάε και έχει ζει το λόγο ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν. Θέλω να σας αναφέρω μια σκέψη μου σύντομα. Αν δεν δούμε τα πράγματα από την προπτική των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών και τη δυνατότητά τους να δράσουν στην ψηφιακή αγορά, τότε χάνουμε διπλά. Γιατί χάνουμε το ψηφιακό εμπόριο και την εσωτερική αγορά, αλλά βέβαια και τα έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί αν έχετε ένα περίπλοκο σύστημα δεν μπορείτε εσείς να αντιμετωπίσετε τις απάτες και αν το σύστημα είναι πολύ περίπλοκο εκείνοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Επειδή είναι περίπλοκο το σύστημα ακριβώ. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να έχουμε μια προσέγγιση η οποία να μας ελευθερώσει από πολλά από τα προβλήματα τα οποία σήμερα αποτελούν εμπόδιο για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις για να εισέλθουν στην αγορά. Θέλω δηλαδή εδώ με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσω τα όσα προτείνονται. Πολλοί το έχουν δει, εντοπίσει το πρόβλημα, αλλά δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Θέλουμε ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά και δεν θα την έχουμε αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απατήσεις του συστήματος ΦΠΑ. Απλοποίηση λοιπόν, απλοποίηση, απλοποίηση για το ψηφιακό εμπόριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η υπερβάνωση Μπερές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή για να ακούσω την παρουσίαση της έκθεσής σας. Τη διάβασα όμως. Διάβασα όλες τις παραγράφους της. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη μου είναι ότι το θέμα αυτό δυστυχώς δεν είναι νέο. Διακυδεύεται η ιστορία αυτή της φοροπάτης για το ΦΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε εξετάσει ξανά στο παρελθόν. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βλέπουμε μια βούληση να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό ζήτημα όπως επίσης να τα βάλει με την φοροποφυγή και τη φοροδιαφυγή γενικότερα όπου αυτή εμφανίζεται. Πρέπει να την υποστηρίξουμε προς την κατεύθυνση αυτή, πράγματι. Όμως δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε παρά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί να τα παίρνουμε από το ένα χέρι και να τα βάζουμε στο άλλο. Δηλαδή, εδώ δεν πρέπει να καταστρέψουμε αυτό το οποίο αποτελεί και την δύναμη της εσωτερικής μας αγοράς. Έχοντας αυτό υπόψη, λοιπόν, έχω να κάνω τις τρεις μου παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την προσαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στην σύγχρονη οικονομία, στον ψηφιακό κόσμο, στην αναγκαιότητα να έχουμε μικρές ενιές ε, θηρίδες, νομίζω ότι όλα αυτά πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερη παρατήρηση. Αν στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πάση θυσία, δεν συνηθίζεται, αλλά εδώ θα ε, συμφωνήσω με τον κύριο Χοκμάρ. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Και όσοι θέλουν ε, πειραματικό πρόγραμμα βάσει του οποίου το βάρος της ευθύνης θα πέσει στον τελικό λιανικό πολιτή, αντιβαίνει στο πνεύμα της εσωτερικής αγοράς, αλλά και στις συστάσεις του πέψε του ΟΣΑ, ενώ εμείς τις θέλουμε και συμφωνούμε με αυτές. Συνεπώς προσοχή. Δεν μπορούμε να ξεκάνουμε ό,τι έχουμε μέχρι τώρα και να επανέλθουμε σε μια εθνική λογική. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που αναφέρονται στις προτάσεις της Επιτροπής για να αντιμετωπιστεί αυτού του είδους η απάτη και αυτούς θα πρέπει να προτιμήσουμε αντί να ξεκάνουμε μία βάση της εσωτερικής αγοράς. Και έρχομαι τέλος και στα ποσοστά ΦΠΑ. Εδώ χρειάζεται πράγματι ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τρευλώσεις ανταγωνισμού που εισάγονται εξαιτίας διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ σήμερα. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε στο παράθυμο όσο έχει σήμερα. Τέλος, ο εισηγητής θα καταλάβει ότι συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 28 της πρότασής του. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Ραπώνη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, παρόλο που οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα δράσης έχει κυρίως στόχο να πετύχουμε από πλευρά του Συμβουλίου σαφείς συστάσεις. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζονται διάφορα ζητήματα. Η καταπολέμηση της απάτης με συμβατικά μέτρα και εδώ η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών γιατί δεν λειτουργεί καλά επί του παρόντος. Η έκθεση του λεκτικού συνεδρίου το λέει σαφώς ότι πρέπει να ενισχυθεί και η αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών και να ενισχυθεί και η εθελούσια συμμόρφωση, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα στους υπόχρεους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Αυτά περί διοικητικής συνεργασίας και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή. Έρχομαι τώρα στο σύστημα ΦΠΑ, το οριστικό. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε όλες τις δυνατές λύσεις. Ξεκινήσαμε από 12 δυνατέ ε, λύσεις εναλλακτικέ και αφού τις εξετάσαμε με τις χώρες μέλη και με τους οικονομικούς φορείς καταλήξαμε σε πέντε εφικτές λύσεις. Αυτές οι πέντε λύσεις εξετάστηκαν από εξωτερικούς συμβούλους και βάσει της μελέτης η οποία υπάρχει στο site της Γενικής Διεύθυνσης Ταξιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταλήξει σε μία λύση που είναι εκείνη της φορολόγησης των διακοινωτικών συναλλαγών. Και γιατί κατέληξε σε αυτή τη λύση η Επιτροπή. Γιατί επιτρέπει έτσι να μειωθεί η απάτη στο ΦΠΑ κατά 40 δις, 40% δηλαδή. Και γι' αυτό διάλεξε η Επιτροπή αυτή τη λύση. Η εφαρμογή τώρα της αντιστροφής του βάρους όσον αφορά τις διακοινωτικές ε, συναλλαγές δεν οδηγεί στην ίδια λύση. Γι' αυτό και δεν συμφωνήσαμε με τη λύση αυτή της αντιστροφής της επιβάρυνσης. Για τις ε, ενδοκινοτικές και εσωτερικές ε, τώρα συναλλαγές. Η αντιστροφή της επιβάρυνσης τρευλώνει τη Γενική Αρχή του ΦΠΑ που είναι η κατακαιρματισμένη πληρωμή όπως υπενθύμησε και ένας Ευρωβουλευτής, το BEPS λέει με σαφήνεια ότι πρέπει να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος ΦΠΑ, δηλαδή τις, ε, σε κομμάτια πληρωμής του ΦΠΑ. Όλες οι χώρες εφαρμόζουν το κλασικό σύστημα ΦΠΑ εκτός από μία που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα άλλο σύστημα, sales tax όπως το λένε, που θυμίζει πολύ την αντιστροφή της επιβάρυνσης. Και τι διαπιστώνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες? Το ανώτερο ποσοστό είναι 89%. Σύμφωνα με το Εθνές Ομισματικό Ταμείο, το... ο μέσος όρος της απάτης είναι 30%. Με 27% λοιπόν ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι ελοχεύουν αν εφαρμόσαμε το σύστημα της αντιστροφής της επιβάρυνσης. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική. Αλλά το επαναλαμβάνω, έχουμε ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ. Το άρθρο 113 της Εθνικής μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε με περισσότερη εναρμόνιση και όχι λιγότερη. Το γεγονός ότι δίνουμε εξαίρεση σε δύο χώρες μέλη θα οδηγούσε σε ένα θεμελιώδη ζήτημα. Συνάδει με τη συνθήκη το να συνεχίσουμε με την εναρμόνιση αν έχουμε διαφορετικά συστήματα ΦΠΑ στις διάφορες χώρες μας. Επίσης, η χώρα που θα ήθελε στο εσωτερικό της να εφαρμόσει την αντιστροφή της επιβάρυνσης προτείνει ένα όριο για τα τιμολόγια πάνω από 10.000 ευρώ. Δηλαδή θα έχουμε δύο συστήματα ΦΠΑ μέσα σε μία και μόνο χώρα. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι υπάρχουν απάτη μέσα σε μία χώρα μέλο και μόνο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική και προσπαθεί να εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα και τους κινδύνους για τις άλλες χώρες μέλη. Γιατί αν επιτρέψουμε εξαίρεση για μία χώρα μέλος, είναι πολύ πιθανόν τα προϊόντα τα οποία δεν φορολογούνται να καταλήξουν σε μία άλλη χώρα. Και αν το ΦΠΑ τον εισπράξουμε στο τελευταίο στάδιο της, ε, στην τελική κατανάλωση δηλαδή, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για ορισμένες χώρες αν μη τι άλλο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική πριν ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ή είναι εναρμόνιση το να προσφέρουμε εξαιρέσει σε τόσο σημαντικές αρχές και αυτό είναι θεμελιώδες. Αν λοιπόν το πειραματικό σχέδιο ήταν το πρώτο στάδιο για ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ το οποίο θα βασίζεται σε ένα σύστημα αυτό της ρευστοποίησης, ιδίας ρευστοποίησης, τότε καταλαβαίνετε ότι η αρχή αυτή δεν μπορεί να δουλέψει. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας το σύστημα του ΦΠΑ που λέμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα 20 χρόνια, δεν είναι αλήθεια. Η τελευταία μας ανακοίνωση ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στην Πράσινη Βίβλο και προηγουμένως είχαμε κάνει και άλλες ανακοινώσεις. Θέλαμε να απλοποιήσουμε τις διατυπώσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα δράσης μας και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε όλα τα αρνητικά στοιχεία του Mini One Stop Shop, να το διευρύνουμε δηλαδή αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, αν μη τι άλλο, κάποιες εξαιρέσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά όλα υπάρχουν στο πρόγραμμα δράση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραπόνιλο Πρόεδρος. Ο εισηγητής τώρα. Τελευταίες σας παρατηρήσεις γι' αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, βλέπετε τη συζήτηση πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να πω πως ο κύριος Ραπόνι έχει δίκιο. Δεν οφείλεται στην Κομισιόν το ότι δεν είχαμε πρόοδο, αλλά στο ότι τα κράτη-μέλη δεν το ήθελαν και αυτό χρεώνεται στην αρχή της ομοφωνίας. Γι' αυτό ήταν η πρότασή μου, κύριε Λούκε, στην οδηγία πλαίσιο, όχι στο ύψος του ΦΠΑ. Εκεί πέρα υπάρχει εθνική αρμοδιότητα. Στην οδηγία πλαίσιο, στην νομοθετική διαδικασία να υπάρξει πλειοψηφία. Και μην ξεχνάμε πως ε, είχαμε πει για ε, ελάχιστο και μέγιστο ΦΠΑ 15 και 25% ε, το 25 δεν πέρασε και είχαμε μιλήσει με τους Υπουργούς Οικονομικών και τότε η Γερμανία και η Γαλλία είχαν πει πως θα πρέπει να υπάρχει τακτική νομοθετική διαδικασία μόνο για το πλαίσιο, την οδηγία πλαίσιο, όχι για το ύψος. Οπότε πράγματι δεν οφείλεται στην Κομισιόν. Για τις ε, ε θα αναφερθώ για τις τοποθετήσω συναδέλφου, θα αναφερθώ τώρα σημαντικότερα σημεία. Ο μειωσμένος, ο μειωμένος ΦΠΑ. Πράγματι, κυρία Φερέρα, τι να πω, στην Πορτογαλία είναι μεταξύ 6 και 23%. Στη Γερμανία μεταξύ 7 και 19. Στη Γαλλία 4, 10 και 21. Στη Μεγάλη Βρετανία 0, 5 και 20%. Οπότε Επίσης, το ποια πράγματα υπάγονται στο μειωμένο ΦΠΑ. Μπορούμε να το δούμε από το πρίσμα της δικαιοσύνης των κάποιων βασικών αγαθών, αλλά εάν υπήρχε ένα ενιαίο πλαίσιο νομίζω πως θα ήταν πρόοδος. Αλλά ε, η Κομισιόν θέλει να τα αφήσει τελείως ελεύθερο στα κράτη-μέλη. Δεύτερο, η καταπολέμηση της απάτης. Εδώ πέρα συμφωνούμε. Και όσον αφορά τη διαδικασία της αντίστροφης χρέωσης, υπάρχει ήδη στη στο διασυνοριακό εμπόριο αυτό το οποίο πρότεινε ο συνάδελφος από τους πράσινους για να μείνουν ε, ελεύθερα τα κράτη-μέλη για να κανονίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε. και θεωρώ πως η σημερινή τεχνολογία και η συνεργασία των κρατών μελών μπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ την κατάσταση. μα. μια συζήτηση με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είχε πει πως ε, αυξήσαμε δραματικά τα έσοδα του ΦΠΑ από όταν ε, περάσαμε τις αυτόματες ταμιακές μηχανές δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ναι, ναι, υπάρχουν διαφορές, πράγματι. Ε, μπορεί να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη. Μετά. Έχουμε το θέμα του ποιες ε, λύσεις έχουν εξεταστεί εδώ πέρα. Είπαμε πως η μεγάλη αυτή επιστημονική μελέτη εξετάζει πέντε εναλλακτικέ. Είναι στατικά όμως αυτά, δεν είναι δυναμικά και μπορούμε να το συζητήσουμε από επιστημονική σκοπιά, αλλά η Κομισιόν είπε ότι ε, θέλει να καταπολεμήσει μόνο την απάτη καρουσέλ αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα ζητήματα τα αφήνουμε στα κράτη-μέλη. Και η εμπειρία μου είναι, μετά από 20 χρόνια στο Κοινοβούλιο, και όπως σωστά είπατε, το πρόβλημα είναι στο Συμβούλιο. Καλό θα ήταν να γίνει μια δημόσια συζήτηση και να έχει και μια συναπόφαση το Κοινοβούλιο. Για το πλαίσιο, όχι τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Βεβαίω, εντάξει, αν θα βρει τώρα πλειοψηφία είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ε, κάνουμε προτάσεις και ας μην τις ε, ψηφίσει η πλειοψηφία και πέρα από το χρονοδιάγραμμα εγώ θεωρώ πως πρέπει να γίνει και μια ακρόαση για αυτό το θέμα κύριε Πρόεδρε δεν γίνανε πριν τις διακοπές γιατί η Κομισιόν είπε πως ε, θα κάνει για τις μικρομισίες επιχειρήσεις ε, μια νέα πρόταση το 2017 Οπότε μπορεί το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο να κάνουμε μια ακρόαση με ειδικούς. Αυτή θα ήταν η δική μου πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση πράγματι αυτού του σημερινού είναι καλή. Θα το, θα το μελετήσουμε θα το συζητήσουμε με συντονιστέ και τον εισηγητή. Ευχαριστούμε για την πρόταση. Εγώ είμαι υπέρ. Σα ευχαριστώ όλου αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ήταν ε, πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και τώρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Το σημείο 7 αλλά και το 8. Calendar of report. θα πρέπει να δούμε πρώτα το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση Langen. Deadline for Τροπολογίες μέχρι τις 31 Πέμπτου το μεσημέρι. Θα γίνει συζήτηση στις 27 εκτελείες τροπολογίες και θα γίνει ψήφιση εδώ ε, στις 30. Ε, και στην Ολομέλεια θα κατέβει το θέμα την 1η Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι τώρα πάμε στα σημεία 7 και 8. Θα ζητηθούν από κοινού κοινοί κανόνες για τιτλοποίηση. Θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση. Και απαιτήσει πολιτική υποπτία για πιστοτικά ιδρύματα και επιχειρήσει επενδύσεων. Οι εισηγητέ είναι ο Πολ Τάνγκ και ο Παύλο Θάλμπα. Του ευχαριστώ γιατί τα έγγραφά του είναι πλήρη και μεστά και ευθύ αμέσω θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τάνγκ. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τέλος ξεκινά η συζήτηση. Ευχαριστώ τον Μακ Λούις, γιατί είχαμε περίπλοκα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε και ε, ξέρετε υπάρχει και αυτό το έργο και βιβλίο το Big Short οπότε θα σήμερα ζητήσουμε αυτό το καυτό θέμα Οπωσδήποτε και η τιτλοποίηση έχει μακρά διαδρομή και στις ε, είπα η... τότε λέγανε εκεί αξιολόγηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμιά πτώχευσης και τελικά κατέληξαν στο ότι έχει 60% πιθανότητα. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύονται οι άσχετοι κατά κάποιο τρόπο επενδυτές, ε, πώς δεν θα έχουμε κάποια τοξικά αξιόγραφα. Θυμάστε πού κατέληξε αυτή η υπόθεση και πώς τελικά διασώθηκαν τόσες τράπεζες στην Ευρώπη με τα χρήματα των φορολογουμένων. Άρα οποιαδήποτε πρόταση για να αλλάξει αυτή η αγορά των αξιογράφων στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, αυτή την εμπειρία. Άρα, τι μαθήματα αντλήσαμε από το παρελθόν και από τα σφάλματα που έγιναν. Ακριβώς εζήγησα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την τιτλοποίηση, είχαμε και έργο της εβδομάδας και ε, είπαμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο και θα πρέπει να εξασφαλίσει το Κοινοβούλιο ότι τα μαθήματα του παρελθόντος θα υλοποιηθούν. Άρα θα πρέπει να γίνει συζήτηση και θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόταση και θα πρέπει ομένως να γεφυρώσουμε τις δύο πλευρές. Μερικοί βλέπουν ε, τις ε, ως ε, ευκαιρία. Και όμως από την άλλη μεριά είναι κάποιοι που φοβούνται ότι η κρίση θα ξαναχτυπήσει. Έχουμε 83 οικονομολόγους που χθες είπαν ότι προβληματίζονται και ανησυχούν. Θα πρέπει να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές και θα πρέπει ε, να έχουμε αυτό το STS αυτού του είδους την τίτλοποίηση απλή, διάφανη κλπ. Και ταυτόχρονα βέβαια να δούμε και πώς θα συνδυαστεί με τον ε, κανονισμό CRR αυτών των πιστώσεων. Να γίνει ασφαλέστερη αγορά και να γίνει και πιο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα. Να προσθέτουν τις ΜΜΕ και άρα με αυτή την τιτλοποίηση οι τράπεζες θα μπορούν να μετακυλήσουν ε, τους ε, κινδύνους ε, και έτσι θα υπάρξει ένα σύστημα πιο στεγανό. Να δούμε τι γίνεται με τη μακροπρόθεσμη δανειοδότηση και τι γίνεται με το maturity transformation, τη μετατροπή κατά τη λήξη. Αυτά είναι βέβαια θεωρίες στην πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι σε κάθε αγορά υπάρχουν ασυμμετρίες. Θα πρέπει να γιατρευτεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης, η τιτλοποίηση οδηγεί σε διασύνδεση του χρηματοοικονομικού τομέα και θα πρέπει κανείς να μπορεί να ξέρει από πού προέρχονται οι κίνδυνοι. Υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος Γι' αυτό και χρειάζεται διαφάνεια. Χρειάζονται υποπτικές αρχές, χρειάζεται ξεκαθάρισμα του ποιοι φέρνουν την ευθύνη. Η πρόταση της ε, Επιτροπής προβλέπει συγκεκριμένα διαβήματα, αλλά έχουμε κάποια έγγραφα εργασίας με προτάσεις που επιδέχονται βελτιώσεις. Όπως ένα δημόσιο αποθετήριο για την τυπλοποίηση, όπως καλύτερες δομές της εποπτείας, γιατί χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο οι πολιτικές αρχές τι ευθύνες έχουν. Πάντως θα πρέπει να δούμε δύο θέματα τα οποία δεν φωτίζονται αρκετά από αυτά τα εγγραφά εργασία. Πρώτα πρώτα αυτό το 5% το retention rate και το ζήτημα είναι ότι αυτό αρκεί για να καλύψει τα συμφέροντα των εμπλεκομένων στην αγορά, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτό είναι πολύ υψηλό. Επίσης, άλλο δύσκολο θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα αποκτήσει περισσότερη σταθερότητα και ότι θα έχουμε πραγματικά διαφοροποίηση και ότι θα έχουμε πραγματική ε, διαφάνεια στις ε, συναλλαγές. Άρα μια τυπλοποίηση που να πιάνει τόπο και να αποδίδει και τις δύσκολες ώρες και σε περιόδους καλές για την οικονομία. Εδώ θα βάλω τελεία, Πρόεδρε, και περιμένω πώς και πώς να γίνει η συζήτηση και να ακούσω και τη γνώμη των συναδέλφων. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Εισηγητά. Και τώρα το, το εισηγητή, του Νότμαρ Μαρκάρας για το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε και εισηγητά, σας ευχαριστώ για την πρότασή σας αγαπητέ Πάμπλο. Η πρόταση αυτή λοιπόν για την τυπλοποίηση ε, υπευλήθη το Σεπτέμβριο του 2015 από την Κομισιόν και δημοσιεύτηκε. Και τη συζητάμε πρώτη φορά σήμερα. Βεβαίω ο κόσμος δεν έχει μείνει ακίνητος όταν προσφέρουμε αυτά τα μέσα στους επενδυτές, ε, όταν δεν τα προσφέρουμε, ε, θα στραφούν αλλού ή θα περιμένουν. Ε, οπότε εγώ θα ήθελα να επιμείνω ταχύτητα αν καθυστερήσουμε κι άλλο θα έχουν προβλήματα όσοι θέλουν να βρουν πίστη για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή για οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματική οικονομία δηλαδή. Επίσης, στον πρώτο γύρο θα πρέπει να συζητήσουμε ποια μαθήματα έχουμε αντλήσει από το παρελθόν, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά η ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποίησης είναι πολύ πιο εύρωστη από την αμερικανική από την άλλη. Χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ε, δεν έχουμε σοβαρή ανάκαμψη. Δεν συγκρίνεται με την ανάκαμψη των Αμερικανών, παρά το ότι η δικιά μας αγορά είναι πιο εύρωστη και για να απαντηθεί άρα αυτό το θέμα θα πρέπει ακριβώς να δούμε τις νέες προτάσεις του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Προς το πρόβλημα της ε, σύμμετρης πληροφόρησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε, αλλά η απάντησή μας μπορεί να είναι μόνο μία. Σαφείς κανόνες και μέγιστη διαφάνεια. Χρειάζονται ξεκάθαρα κριτήρια όσον αφορά τους κανόνες για διπλοποίηση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Επιπλέον πρέπει να γίνει μια έντονη συζήτηση για μια ερμηνεία των κριτηρίων και μια ρεαλιστική λύση για την... πώς θα ποινικοποιηθούν οι παραβάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν νομοθεσία χωρίς να ορίσουμε ποιοι είναι οι φορείς ε, και ποιες είναι οι κυρώσεις. Καταλαβαίνετε πως νομοθεσία χωρίς ε, κυρώσεις δεν έχει νόημα και ουσία. Είναι καλό το ότι ε, θέλει ο εισηγητής να θέσει κάποια θέματα στο πλαίσιο των εθνικών κρατών ε, και θα πρέπει για τις εναλλεκτικές λύσεις νομίζω να περιμένουμε την ακρόαση. Και αναμένω λοιπόν προσεχώς το έγγραφο εργασίας να γίνει μια πραγματική έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάρας. Τώρα, εκ μέρους του ECR Messenger. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω προκαταρτικά ότι ανησυχώ λίγο για το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για την έκθεση αυτή. Οι χώρες μέλη στο Συμβούλιο φαίνεται ότι καταλήγουν σε συνένεση και σε 7 εβδομάδες εδώ αναβάλουμε ξανά και ξανά μια αναγκαία νομοθετική ρύθμιση. Αυτή ήταν η προκατακτική μου παρατήρηση. Το Συμβούλιο έχει ήδη πετύχει πολλά. Έχει βελτιώσει κατά πολύ την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς όπου πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο. Πρώτον, όσον αφορά την ε, ευκρίνεια και τη σαφήνεια, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες γιατί είναι πιο ξεκάθαρο το ποια είναι τα κριτήρια του STS της πρωτοβουλίας αυτής απλοποίησης, διαφάνειας και τυποποίησης. Αν μη τι άλλο, όπου τίθενται ζητήματα και κάποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρούνονται στα κριτήρια ασφάλειας της τυποποίησης. Πάντω έτσι καλώς έχει βελτιωθεί όπως είπα το κείμενο τη Επιτροπής από το Συμβούλιο, αλλά εγώ βλέπω και άλλα περιθώρια βελτίωση. Ένα άλλο τομέα που θα έπρεπε να βελτιωθεί πιστεύω γιατί έχει να κάνει με μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ατομικούς επενδυτές έτσι όπως έχει το κείμενο σήμερα βλέπω ότι σε πολλές περιπτώσεις προγραμμάτων ε, ιδιωτικών χρογράφων καλυμμένων με στοιχεία ενεργητικού, το ABCP, θα πρέπει να συμμορφώνονται και αυτά στις προδιαγραφές STS. Κατά συμφωνώ με τα επιχειρήματα και των επενδυτών και του κλάδου που λένε ότι πολλές φορές χρειάζεται ένας τρίτος να εμπλακεί για να κινεί η αγορά, αλλά καταλαβαίνω επίσης και τόσο αναφέρονται το αφορά τον ηθικό κίνδυνο. προκειμένου να υπάρχει αυτή η πιστοποίηση που να μην είναι αυτοπιστοποίηση αλλά να είναι από τρίτο μέρος. Νομίζω ότι αυτό θέλει η ομάδα μου. Όσον αφορά το δημόσιο μητρό, εγώ δεν βλέπω γιατί να πρέπει να υπάρχει κάτι καινούριο για τι τιτλοποίησεις STS. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να υπάρξει μια τέτοια νέα αρχή τη στιγμή που προτείνει ενημέρωση προς τους επενδυτές η Κομισιόν και νομίζω ότι αυτό φτάνει. Υπάρχουν λοιπόν τομείς όπου πρέπει να διορθώσουμε το κείμενο και το θέμα της τρίτης χώρας βέβαια και θα ήταν κρίμα να παρετηθούμε από επενδυτές και εκδότες από τρίτες χώρες και να περιοριστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Έτσι περιορίζουμε την αγορά. Και όσον αφορά για τις τετλοποίησεις που δεν εμπίπτουν στο STS, πρέπει να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίζουμε και αυτές. Τι θα ισχύει για τις τετλοποίησεις μη STS. Δημιουργούμε μια αγορά δύο ταχυτήτων και οι τιτλοποίησεις που δεν είναι STS δεν πρέπει να παραλύσουν. Συμφωνώ πάντως ότι το σημαντικό είναι ο κίνδυνος, γιατί έτσι κι αλλιώς η δανειοδότηση ελοχεύει κινδύνους. Αλλά τι γίνεται όταν δεν τηρούνται τα κριτήρια STS. Είναι πολλά ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα καλά, τα οποία όντω τα αντιμετωπίζουμε στο έγγραφο αυτό και πολύ θα ήθελα το έγγραφο αυτό να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Α, προηγουμένω η Άλτε, ο Πίτερ Γιέστερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η υψηλή ποιότητα τυλοποίηση μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Άρα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση σε κεφάλαιες επενδύσεις, άρα πρέπει να βοηθήσουμε τις τιτλοποίησεις. Πρέπει να δώσουμε όμως πολύ προσοχή στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ABCP τιτλοποίηση, τα χρεόγραφα τα καλυμμένα με στοιχεία ενεργητικού. Να υπάρχουν ε, λοιπόν τα κριτήρια STS, να υπάρχει επιστοποίηση και προβλέψεις για τρίτες χώρες. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια ισχυρή βάση και νομίζω ότι το Συμβούλιο όντω έχει βελτιώσει πολλούς τομείς της εξαιρέσεις, για παράδειγμα, όσον αφορά τα επίπεδα ε, λεκτικότητας, τα θέματα της τιτλοποίησης ABCP και ε, τα θέματα των ε, μεταβατικών προδιαγραφών. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, καλό είναι που ακούμε ότι συμφώνησαν οι συγκητές μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλύτερα αν είχαν συμφωνήσει σε ένα πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Στην ε, ομάδα έχουμε απογοητευτεί από την έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ακριβώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο νωρίτερα. Δεν βλέπουμε καμία σχέση ούτε άμεση ούτε έμεση του STS με την Κεφαλιακή Ένωση. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και για την οικονομία αλλά και γενικότερα. Ο τύπος είδατε ότι αρνητικά το κάλυψε και δυστυχώς δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου. Πάντως ευχαριστώ τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας και προσβλέπω στο σχέδιο έκθεσης και να συνεργαστούμε μαζί του και με τους υπόλοιπους και όδες εισηγητές για το καλύτερο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέει κύριε για τους πρασίνους. Ήδη Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν συμφωνήσει, οπότε απευθύνονται τώρα σε εμά και θέλουν απλώ να δώσουμε το πράσινο φως. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το χρονοδιάγραμμα, αλλά είπαμε ότι ε, ακριβώς η τετλοποίηση ήταν ε, πηγή τη καταστροφή του 2008 και θέλουμε να επαναληφθεί. επομένω θα πρέπει τώρα να κάνουμε τη δουλειά μα σωστά και να την κάνουμε το σωστό timing. επομένω ερωτώ Ποιο ωφελείται εάν γίνει γρήγορα αυτή η συμφωνία στο να το μας λένε ότι θα βοηθήσουμε την ε, ανάκαμψη, θα χρηματοδοτηθούν οι ΜΜΕ, αλλά είναι αυτό μια αυθεντική λύση για το πρόβλημά μα. Πού είναι τα στοιχεία ότι εάν έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, τιτλοποίηση θα βοηθήσουμε τις ΜΜΕ γιατί η δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κοινή προσπάθεια σε επίπεδο οικονομικό, δημοσιονομικό. Έχουμε ε, αυτές όλες τις περικοπές, έχουμε τη λιτότητα. Αυτό πνίγει τις οικονομίες της Ευρώπης. Επίσης, οι ίδιες οι ΜΜΕ δεν θεωρούν ότι αυτά που λέμε εδώ τους λύνει το πρόβλημα. Και η Κεντρική Τράπεζα επίσης θεωρεί ότι η πρόσβαση σε δανεισμό ε, είναι το μικρότερο πρόβλημα των ΜΜΕ. Ε, το 25% οι περισσότεροι πάντων είπαν ότι δεν είναι το δάνειο το πρόβλημα από την ΜΜΕ, αλλά είπαν ότι το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν πελάτες. Εμείς ε, λέμε ότι δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στις πιέσεις για τέτοιου είδους τιτλοποίηση, θα πρέπει να υπάρξει πάντως ευρεία συνένεση για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους από μια νέα οικονομική κρίση που τελικά οι ίδιοι θα πληρώσουν την ύφη για αυτήν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι τροπολογίε θα κάνουμε για διάφορα ζητήματα όπως ήδη αναφέρθηκε το skin in the game και θα πρέπει να δούμε με τι δυναμητικό πρότυπο θα υπάρχει, να υπάρχει λογική στη δανειοδότηση, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η έκθεση των τραπεζών στον κίνδυνο, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, πριν υπάρχει η τιτλοποίηση, να μπορέσουν να αναχθούν τα δάνεια και έτσι να είναι βιώσιμες οι τράπεζες ή βιώσιμα τα δάνεια. Θα πρέπει επομένω να περιορίσουμε την ε, ε, τιτλοποίηση σε συγκεκριμένα αξιόγραφα και έτσι να μην ε, υπάρχουν κινητές αξίες που είναι τα περίφημα σκουπίδια. Άρα θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός εργαλείων και μέσων. Το θέμα είναι τώρα ποιος θα είναι η ρυθμιστική αρχή, να μην έχουμε μία βιζαντινολογία μην θέλουμε να καλύψουμε με ένα κείμενο πάσα δραστηριότητα να έχουμε το, να μην έχουμε το πρόβλημα το ότι η εξειδικευμένη τιτλοποίηση δεν πιάνει τόπο. Χρειάζεται ειδικό καθεστώς για κάθε προϊόν. Ειδική τιτλοποίηση και επίσης είμαστε κατά του μοντέλου ε, έγκρισης που προτείνεται και αυτή η αυτοπιστοποίηση θα πρέπει να οδηγεί σε απάτες. Χρειάζεται συντονισμός σε επίπεδο εποπτείας. Να αντιμετωπιστούν επομένως οι κίνδυνοι και τα προβλήματα με τη σωστή εποπτεία και ρύθμιση. Επίσης, όσον αφορά τα κατανεμημένα εργαλεία και μέσα, και αυτό είναι πρόβλημα της ε, τιτλοποίησης που είχε ανακύψει την εποχή της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή, πολύ χρήσιμο το έγγραφο θέλουμε να είναι επικοδομητική η συνεργασία μας, να φέρουμε την ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή οικονομία και να μην ε, στηρίξουμε απλώς την ε, κεντρική τράπεζα σε σχέση με την νομισματική πολιτική που θέλει να χαράξει. Ο κύριος Μάρκο Τσάνι είναι εδώ. Όχι. Επομένως, προχωρούμε. Στην έκθεση του κυρίου Παύλο Θάλμπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία από τις προτεραιότητες Η κυρία Μπέρες εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε. Συγγνώμη, το έγγραφο δεν είναι στους φακέλους από ό,τι φαίνεται και ο εισηγητής μου είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα διανεμήθη, αλλά μήπως μόνο του σκιώδης, γιατί εγώ δεν το έχω. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κείμενο σε χαρτί, θα ήταν χρήσιμο. Πρόεδρος Εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους. Αλλά όχι από ό,τι φαίνεται σε χαρτί εξαιτία των νέων κανόνων εξοικονόμησης χάρτου που έχουμε υιοθετήσει με ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο εφόσον το ζητήσετε το έχετε σε χαρτί. Ο κύριος Ζάλου Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν έλεγα ότι μία από τις κύριε προτεραιότητες της θητεία μας αυτή είναι η ενιαία αγορά κεφαλαίων. Και με αυτό έχουν να κάνουν οι δύο εκθέσεις που συζητάμε σήμερα. Και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ενιαία αγορά κεφαλαίων. Πρέπει να εξηγήσουμε ποιε είναι οι πηγέ χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίω, που δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται μόνο με, από τις τράπεζες, αλλά πρέπει να έχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Και ο στόχος είναι ένας, είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναμφίβολα η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, γι' αυτό σήμερα είναι περισσότερο σημαντική παραποτέ η συζήτηση και οι εκθέσεις αυτές που εξετάζουμε σήμερα. Η ενιαία αγορά κεφαλαίων και οι τιτλοποίησεις θα επιτρέψουν να έχουμε πιο ολοκληρωμένες οικονομικές αγορές, πιο ανοιχτές, πιο ανταγωνιστικές και τελικά πιο αποτελεσματικέ. Είμαστε μπροστά σε μια ιστορική σημασία στιγμή για να προχωρήσουμε προς την δεύτερη αγορά κεφαλαίων και προκειμένου να το πετύχουμε αυτό είναι αναγκαίο να συζητήσουμε και να κρίνουμε τις δύο αυτές εκθέσεις που όπως ε, είπα συζητάμε σήμερα. Είχαμε οικονομικές κρίσεις. Είχαμε πριν μια αγορά τιτλοποίησεων που λειτουργούσε καλά και μάλιστα οι αγορές αυτές είχαν και μια σχετικά ικανοποιητική αντίδραση στις οικονομικές κρίσεις που ζήσαμε. Τώρα οι νέες προδιαγραφές, οι νέες οικονομικές προδιαγραφές όπου εγκρίνουμε σιγά σιγά, όπως επίσης και το περίφημο στίγμα κατά τον τιτλοποίησεων φρέναρε κάπως την ανάπτυξή τους. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σχετικά με αυτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία λοιπόν ότι αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ και αν καταφέρουμε να γίνει πραγματικότητα, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για τους επενδυτές, θα ήταν μια ευκαιρία για να βελτιωθεί η λειτουργία των κεφαλαικών αγορών, θα ήταν μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε επίσης και την τοποθέτηση των πόρων. Θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις, θα διαφοροποιήσουμε και τις πηγές χρηματοδότησης και τελικά θα είναι και μια ευκαιρία προκειμένου να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, επιμένω, ότι πρέπει να πετύχουμε την ολοκλήρωση των κεφαλαικών αγορών και να διαφοροποιήσουμε, όπως είπα, τις πηγές χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να πετύχουμε οι ε, δημοσιονομικές, ε, δημοσιονομικοί φορείς και παράγοντες να μπορούν να διευκολύνουν την χρηματοδότηση και να ενισχύσουν την χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία κατά τη γνώμη μου σχετικά με τα οποία πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο στην έκθεση αυτή. Το ένα είναι η προτεραιότητα εκτίμηση, off approaches όπως λέμε στα αγγλικά. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις. Είδαμε πρώτα απ' όλα την πρόταση της Επιτροπής, είδαμε την πρόταση του Συμβουλίου, είδαμε εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχουμε και την πρόταση επίσης της ε, Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Όλα αυτά είναι στοιχείο κλειδί της έκθεσης αυτής και γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη των σχεδόν εισηγητών αλλά και των υπολείπων συναδέρφων. Χωρίς καμιά αμφιβολία αυτό είναι και το πιο ευαίσθητο κομμάτι της έκθεσης. Κατά τη γνώμη μου, απόλυτη προτεραιότητα, προτεραιότητα είναι η τιτλοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται να διευκολύνουμε όταν θα έχουν εγκριθεί όλες αυτές οι εκθήσεις τις τιτλοποίησεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αναμφίβολα αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι μπορούμε να τον πετύχουμε αυτόν τον στόχο και μάλιστα χωρίς να διακινδυνεύσουμε με την δημοσιονομική σταθερότητα που σίγουρα αποτελεί και αυτή μια βασική μας προτεραιότητα δίχως άλλο και των δύο αυτών εκθέσεων. Όπως ακούσαμε φυσικά και υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο εκθέσεις και χωρίς καμιά αμφιβολία και οι δύο συγητές όπως οι σκιώδεις οι συγητές έχουμε δεσμευτεί να συντονίσουμε το έργο μας γιατί δίχως άλλο αυτό θα αποβεί σε όφελος όλων. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε και ο Βολτάν, υπάρχει μια συμφωνία επ' αυτού μα να με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά αν υπάρχει συμφωνία να επιταχύνουμε κάπως το ρυθμό μας, δεν έχω αντίρρηση. Πρέπει να υπάρχει συνένεση όμως. Αυτά. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω να μπορέσουμε να δουλέψουμε επικοδομητικά μεταξύ μας και σύντομα να διαπιστώσουμε ότι ο κοινό μας στόχο που είναι η ανάπτυξη και απασχόληση θα υλοποιηθούν χάρη ακριβώ και στις εκθέσεις που συζητάμε σήμερα. σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος ε, Φερνάντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα, πρώτα, να ευχαριστήσω για το έργο το οποίο επετέλεσε ο εισηγητής και όλους όσους τον ε, βοήθησαν για να επεξεργαστούμε ε, τον ορισμό αυτών των νέων τιτλοποιήσεων που θέλουμε να είναι τυποποιημένες και με διαφάνεια και έτσι να μπορέσουμε να τονώσουμε την ε, κεφαλαία αγορά όπως τόνισαν και οι προλαλήσαντες για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτής της κεφαλαία αγοράς εμείς οι σοσιαλιστές Θέλουμε να εξεταστεί το πώς θα τονωθεί η κεφαλή αγορά και η προσέγγιση μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσοχή γιατί έχω το 2007 και μετά είχαμε πολλά προβλήματα όσον αφορά την ευθυγράμμιση ε, ε, των κερδών και του ρίσκου. Ε, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρα και αυτό ε, είναι μία από τις αιτίες της σημερινής ε, κρίσης. Και στις ε, είπα προέκυψε αυτή η δυσκολία. Δεν μπόρεσε το κέρδος να ευθυγραμμιστεί με το ρίσκο για αυτά τα προϊόντα, για αυτές τις κινητές αξίες. Οπότε και θα πρέπει να δούμε πώς θα περιχαρακώσουμε τον ορισμό της τυπλοποίησης αυτής. Να συζητηθεί αυτή η πρόταση ούτως ώστε να δούμε ποιες είναι οι κεφαλαιοχικές απαιτήσει που σχετίζονται με αυτές τις τιτλοποιήσεις, να δούμε πώς θα μπορέσουμε τα πράγματα να είναι πιο απλά, πιο ελαφρά για αυτή την ε, κεφαλαιοχική απέτηση. Άρα μεγάλη προσοχή. Και άρα θα πρέπει να είναι πολύ στεγανός ο ορισμός των τιτλοποιήσεων και οι δύο εκθέσεις λοιπόν έχουν ε, και είναι πορεία γιατί είπαμε ότι αυτές οι αιστείες, αυτές οι τυλοποίησεις απλές κλπ θα πρέπει να συνοδεύονται από πολύ προσεκτική πρόβλεψη των κεβλουχικών απαιτήσεων και αυτές οι τυλοποίησεις θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πραγματικά απλές, διάφανες και επομένως να υπάρχει μία ρύθμιση φιλόδοξη και όπως είπαμε για την κυβλουγική απέτηση να ενεργήσουμε τρόπο που να ελαφρώσει, να απλουστεύσει τα πράγματα. Και ο απότερος στόχος ε, αυτής της προσπάθειας που είναι στα πλαίσια της ε, ενίας κεφαλαίου αγοράς ακριβώς είναι στο να καταλήξουμε μια τέτοια ολοκλήρωση αυτής. Ε, μας είπε και ο Παύλο για την ιεράρχηση των συστημάτων υπολογισμού αυτών των ε, κεβουαλιστικών απαιτήσεων και έχουμε το θεματολόγιο, το νομοθετικό. Θέλουμε να δούμε το τι θα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, πίεση από τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης και επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την επίλυση αυτού του προβλήματος το οποίο μας προβληματίζει και αυτό γιατί αφού το κρατικό χρέος συνδέεται με τον κίνδυνο των τυπλοποιήσεων τότε θα πρέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση να ενεργήσουμε δηλαδή να φτιάξουμε μια αυθεντική κεφάλαια αγορά στην Ένωση και θα πρέπει επομένως να αποκαταστήσουμε την ορθή ιεράρχηση των ε, κεφαλικών απαιτήσεων. Και ε, βέβαια θα πρέπει αυτό να γίνει με μια απλή και διαφανή τυποποιημένη τιτλοποίηση όπως λέει η έκθεση του Πολ Τάγκ. Επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε, συγκροτώντας δύο ομάδες εργασίας που θα πρέπει να προχωρούν χέρι-χέρι και όχι απομονωμένα. Να είναι ξεκάθαρη αυτή η ευθυγράμμιση για ρίσκο και κέρδη και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Θα πρέπει να ε, προσέξουμε το τι πνεύμα θα διέπει αυτή, αυτή την ε, κοινή κεφαλή αγορά σε σχέση με τις εθνικές κεφαλαίου. Ο κύριος Καμάλη το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συγητές και τους κοιόδη συγητές πρώτα απ' όλα. Πρέπει να πω πώ εδώ δεν ξέρω τι να πω γιατί αφενός αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες για την βραδιτητά, από την άλλη θεωρώ πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Και τι εννοώ. Όπως λέει και ο Πολ και έχουν πει και άλλοι, Έχουμε όντως μάθει τα μαθήματα ε, της κρίσης, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά της τιτλοποίησης. Ακούγοντας την σημερινή συζήτηση βλέπω πως χρησιμοποιούμε ακόμα την ε, γλώσσα που θέλουν αυτοί που προσπαθούν να μας μπερδέψουν. Π.χ. μιλάμε ακόμα για τίτλους ε, οι οποίοι βασίζονται σε κάποια στοιχεία του ενεργητικού. Μα γνωρίζουμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δείτε το τι ήταν αυτά, ήταν ένα ωραίο όνομα για ένα ομόλογο που βασίζονταν σε εργαστικά subprime. Και εξακολουθούμε όμως να χρησιμοποιούμε αυτή την ε, γλώσσα των διεφθαρμένων εκείνων οι οποίοι προσπάθησαν να μας δουλέψουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ασφαλή αγορά Οπότε ναι να πάμε γρηγορότερα, αλλά ταυτόχρονα δεν σημαίνει ταχύτητα ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τα μαθήματα της κρίσης και να μην μας γελάνε, όπως είπα αυτοί οι οποίοι μας δούλεψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όποιος έχει διαβάσει το The Big Short, το Fool's Gold και τα άλλα βιβλία για την κρίση, θα δούμε το πώς ε, ξεγελάστηκαν ε, οι ρυθμιστικές αρχές από ανθρώπους πολύ εξυπνότερους ε, που φρόντιζαν να εκμεταλλεύονται το σύστημα ειδικά όταν μιλάμε για τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Δηλαδή εγώ θέλω να δουλέψει το σύστημα, αλλά να είμαστε και επιφυλακτικοί για αυτά τα οποία μας λέει ο κλάδος. Και συμφωνώ εδώ πέρα με το Μολυριά το επιχείρημα αυτό περί που θα απελευθερώσει κονδύλια για να δώσουν οι τράπεζες λεφτά στις μικρομισές επιχειρήσεις ή μήπως απλά θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά για να αγοράσουν και όχι να λύσουν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε λοιπόν, το πρόβλημα των κεφαλαίων είναι ακριβώ ότι αναζητούμε υποτίθεται εναλλακτικέ από την χρηματοδότηση των τραπεζών. Και εδώ πέρα υπάρχει κάποια αντίφαση ότι θα απελευθερώσουμε δηλαδή κεφάλαιο για να το δανείσουν οι τράπεζες και ελπίζουμε να το δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας πούμε λοιπόν τώρα στις λεπτομέρειες. Ας δούμε παραδείγματο χάρη την ε, ιεραρχία που υπάρχει εδώ πέρα για τον υπολογισμό του πιστοτικού κινδύνου. Μήπως ε, εμπιστευόμαστε πάρα πολύ εδώ πέρα τις υπηρεσίες ε, αξιολόγησης. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τα εσωτερικά της, των τραπεζών. Ποιος θα τα αμφισβητήσει, θα υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν ή θα τους δουλέψουν μετά. Εξωτερικές αξιολογήσεις. Έχουμε ήδη ακούσει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα για τις ε, εταιρείε αξιολόγησης και άρα μένουμε μια τυποποιημένη προσέγγιση για την τιτλοποίηση. Και τι καταλαβαίνουμε από αυτό πράγματι. Και τέλος να φροντίσουμε να έχουμε πραγματικές κεφαλιακές απαιτήσεις και να μην χρησιμοποιούνται εξισώσεις για να εκμεταλλευτούν το σύστημα. Και μην ξεχνάμε το θέμα της ε, IAG, η οποία ε, τελικά είχε εκτεθεί σε κάποια μέσα αξίας 8,2-3 ε, εκατομμυρίων και όταν κατέρευσε δεν είχαν επαρκές κεφάλαιο για να πληρώσουν. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε εμείς να υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ, Σαΐτ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα για τους φιλελεύθερους. Πέτερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν διαβάσω την παρέμβαση του Μάικλ Τόρερ, ο οποίος ε, απουσιάζει, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το χρονοδιάγραμμα. Αλλά, βεβαίως, ε, αργά δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε και σωστά και αντιστρόφως και εδώ πέρα βεβαίω μιλάω εγώ και εκπροσωπώ την ομάδα, όχι τον κλάδο. Λοιπόν, τώρα, τα όσα λέει ο συνάδελφος. Καλώ ορίζω την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για μια απλή και διάφανη τίτλοποίηση η οποία... Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ συνάδελφοι, ξέρω πως έχετε πολλά να συζητήσουν οι πράσινοι και οι κομμουνιστές φίλοι, αλλά ε, φίλοι εντό εισαγωγικών. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ε, θα είπα να ακούσουμε λίγο και τον ε, ομιλητή μας. Στους συμβούλους απευθύνομαι, στους συμβούλους της ομάδας. Εντάξει, μην παρενοχλείτε την συνεδρίαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν. ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αυτό μπορεί να μπορεί να ωφεληθούν, δηλαδή οι τράπεζες να δώσουν περισσότερες πιστώσεις αν έχουν πιο διαφοροποιημένες στρατηγικές χρηματοδότησης. Οπότε μπορεί η τιτλοποίηση αυτή να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να απευθυνθούν στις κεφαλαίες αγορές. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα γιατί η συνθετική τιτλοποίηση αποκλείεται από την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ακούσαμε από πολλές πλευρές πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά θα προτιμούσαν ε, συνθετική τυπλοποίηση. Οπότε ενδιαφέρον θα ήταν η Κομισιόν να μας εξηγήσει γιατί δεν περιλαμβάνονται εδώ πέρα και να δούμε με τους συναδέλφους αν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιτευχθεί αυτό καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός στόχος. Για τα ABCP θα ήθελα να πω πως σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς οι κεφαλαιακές απαιτήσει για κάποιους ε, τύπους τέτοιων προϊόντων και λοιπόν συναλλαγών ABS ε, θα αυξηθούν σημαντικά στην πρόταση της ε, Κομισιόν και στη συμβαστική του Συμβουλίου. Μας παρουσίασαν κάποιους υπολογισμούς με βάση την προσέγγιση του ERBA, παραδείγματος χάρη αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης για ένα γερμανικό αυτοκίνητο παραδείγματος χάρη μέχρι και 250%. Είναι σημαντικό αυτό για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστραφούν από την ομοθεσία όπως αυτή προτείνεται. Αυτό το ζήτημα λοιπόν θα ήθελα να το δούμε. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω την σημασία που αποδίδουμε στην αναζωογόνηση της ε, αγοράς αυτής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο. Εμείς είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι από το Συμβούλιο και οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η πρόοδος ε, στο φάκελο αυτό με την πρόοδο στο ΙΔΙΣ δεν είναι αποδεκτή. Αυτά εξ ονόματος του κυρίου Τόρια. Σας ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Βλέπω οι κομμουνιστές ακόμα κουβεντιάζουν. Μόλι κόρτη για του πρασίνου. Μόλι έχει το λόγο. Σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα θα σα πω ότι άξιζε να έρθω στην συνεδρίαση. Συμφωνούμε με τον συνάδελφο. Είδατε όλα γίνονται, όλα γίνονται. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Δεν έχουν προχωρήσει βέβαια τόσο πολύ, ούτω ώστε να ε, τα ολοκληρώσουμε όσο είχαμε να πούμε οι σκιώδε. Αλλά έχω τι εξή παρατηρήσει βασικά. αυτό τα οποία λέμε είναι πόσο κεφάλαιο κινδύνου θα πρέπει να επενδύουν στην επιστοποίηση, στην τιτλοποίηση οι τράπεζε. Οπότε θα πρέπει έτσι να ε, εξαλαφρώνεται ο ισολογισμό. Και θα πρέπει να δούμε το ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση των ε, τραπεζών. Να πώς ξεπίδησε η κρίση. επομένω αυτό που χρειάζεται είναι προσοχή και επιφύλαξη. Να, πώ ε, αλληλοσυνδέονται οι δύο εκθέσει και εγώ είμαι σκιώδη και για τι δύο. Μόνο εγώ είμαι και για τι, δύο, αλλά προσπαθώ να το αξιοποιήσω σε όλη τη διαδρομή. Και θέλω να σα πω πω εμεί οι πράσινοι τα βλέπουμε πρώτα-πρώτα. Αυτοί οι κανόνες επιφύλαξης τη τράπεζα για την πραγματική οικονομία. Θα είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε περιθώρια περιθώρια διακινδύνευσης στην τράπεζα για να τονώσουμε την οικονομία και να μην υπάρχει <clears throat> επιφύλαξη για τον τραπεζικό τομέα ούτω ώστε δήθεν να βοηθήσουμε την οικονομία γιατί οι πολίτες αγωνιών όποτε εμεί χαλαρώνουμε την προσοχή μας για το τραπεζικό, τον τραπεζικό τομέα και αυξάνει η ανάληψη ρίσκου. Ε, βέβαια υπάρχουν και άλλοι κλάδοι και υπάρχουν και άλλα στοιχεία του ε, ενεργητικού σε σχέση με τα, ε, με τα στεγαστικά τα ταμιευτήρια. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα πρέπει να φτάσουμε σε, σε, σε θέσπιση ορίου για την τιτλοποίηση σε σχέση με το τι καλύπτουν αυτές τις τιτλοποίησεις από πλευράς κεφαλαίου εταιρικού ή στοιχείου ενεργητικού. Δεν βλέπω από το διευθυντή κάποιον. Κύριε Μόνο. Α, μιλάει στο τηλέφωνο. Αλλά η κυρία Μπελέση έχει δείξει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποια στιγμή θα πρέπει πρόεδρε Γκουαλτιέρη να μας πείτε γιατί έχετε επιταχύνει την εξέλιξη σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει ρόλο να διαδραματίσει ούτως ώστε τα πράγματα να προχωρούν με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός στους συμπολίτε. Τιτλοποίηση. Τι είναι αυτά, αυτά είναι ε, κινέζικα. Ε, Securization στα αγγλικά, στα γαλλικά. Μα τι γίνεται. Είδατε τι έγινε στην κρίση. Γιατί επομένως να προχωράμε προς γρήγορη νομοθέτηση χωρίς να έχουμε α, κάποιες ε, στέρες εγγύσεις. δηλαδή τι έγινε και με το Συμβούλιο και αυτοί βιάζονται ούτω ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση των ΜΜΕ που δεν υπάρχει σήμερα. Άρα χρειάζεται, σύμφωνα με το πλάνο Γιούνκερ, να βρεθούν οι καινούργιες πηγές χρηματοδότησης και έτσι να δούμε τι γίνεται με τα non-performing loans. Κάτι σαν κόκκινα δάνεια. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά με την ελόγω πρόταση. Να, ξεκινάω με το πλάνο Juncker. Έγινε προηγουμένω συζήτηση εδώ για την έκθεση Φερνάντες Μπούλμαν και είπαμε ότι η σωστή αφετηρία για υλοποίηση του πλάνου Γιούγκερ είναι να υπάρξουν κρατικά όλα, και να μην εμπιστευτούμε το κλειδί στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε η χρηματοδότηση της οικονομίας θα εξασφαλιστεί με την ανάληψη του κινδύνου, λένε εδώ, από τον ιδιωτικό τομέα. Σχεδόν δίνουμε επιταγή εν λευκό στον ε, ιδιωτικό τομέα. Άρα πέραν της Επιτροπής και εμείς ως Κοινοβουλίο θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει επομένω να θωρακιστεί η υποπτία όπως σωστά είπαν οι συγκητέ. Θα πρέπει να, προσέξουν προσέξουμε επίσης ποιος είναι ο ρόλος των εταιριών ε, αξιολόγησης. Γιατί ξέρουμε τι έγινε και με αυτές στην κρίση. Θα πρέπει επομένως να δούμε πώς θα συνεχιστεί η μακρόπνοη δανειοδότηση. Έτσι θα πρέπει να συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο δημιουργικό, ούτω ώστε ο νομοθέτης να δώσει τη σωστή κατεύθυνση σε αυτήν την ανάκαμψη. Να μην προχωρήσουμε στα τυφλά. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε κατευθύνσει προς τον νομοθέτη. Μιλάμε για μακρόπνες επενδύσεις, μιλάμε για το πλάνο Juncker υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική που εμείς θέλουμε ούτω ώστε να είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Να καλυφθούν και οι οικολογικές μας ανησυχίες και έτσι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την, την... Ε, το πλάνο Γιούγκερ. Είμαστε στην αρχή τη διαδρομή και όχι στο τέλο, λέει ο πρόεδρο. Τέλο πάντων, δευτερολογεί τώρα ο κύριο Τάγκα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πολύ μου άρεσαν αυτά που είπε ο Σέιντ ότι θέλω να εργαστώ, γι' αυτό είμαι σκεπτικής Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δουλέψει κανείς και εδώ στην τυπλοποίηση χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Και για να την πετύχουμε χρειαζόμαστε χρόνο, σκληρή δουλειά θα είμαι σύντομο, όπως είπα. Άκουσα πολλές καλές επικοδομητικές παρατηρήσεις που θα οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα υπάρξουν βελτιώσεις δηλαδή παρετέρω στην πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε. Ο άλλος εισηγητής τώρα, Πάμπλο, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ναι, θα είμαι και εγώ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και όλους τους συναδέρφους που πήραν το λόγο και μας είπαν τη γνώμη τους. Και εγώ λέω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φυσικά είναι σαφές ότι μία από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι οικονομική σταθερότητα. Και μία από τις προτεραιότητες μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι το στοιχείο κλειδί για τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν θα εφαρμοστεί η κεφαλιακή ένωση, τότε θα το δούμε αυτό. Αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό που κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνω και τις ανησυχίες για το ATS ε και όταν συζητάμε για ένα σπιράλι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σίγουρα τα μαθήματα που πήραμε από την κρίση. Όσον αφορά την ιεραρχία της προσέγγισης και τον ρόλο των οργανισμών χρηματοπιστωτικής, αξιολόγησης χρηματοπιστωτικής ικανότητας, σίγουρα θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος τους, τι ρόλο θέλουμε να τους δώσουμε. Επίσης, συμφωνώ με τις ανησυχίες που ακούστηκαν για τον κίνδυνο μετάδοσης και τελικά όλα αυτά θα συνδεθούν με το STS. Διαφάνεια, όπως είπαμε, απλοποίηση. Οπότε, στο τέλος, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα σχόλιά σας και προσβλέπω σε συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε μια ισορροπημένη έκθεση με συνεργασία μεταξύ όλων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την σημαντική αυτή συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δημόσια ακρόαση αρχές Ιουνίου και θα εξετάσουμε στις 21 Ιουνίου την έκθεση και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι 20 Ιουλίου για τη μία έκθεση και 22 Ιουλίου για την άλλη. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει τον Οκτώβριο για να εξεταστούν οι τροπολογίε και τον Νοέμβριο να, εξεταστεί, να εξεταστούν οι εκθέσει εδώ στην ΕΚΟΝ και το Δεκέμβριο να πάνε στην Ολομέλεια. Οι συζητήσει συνεχίζονται, οι συντονιστέ και εγώ ίδιο. Θα το κοιτάξουμε αυτό, μήπω δηλαδή θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε λιγάκι το ρυθμό Από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι συντονιστέ συμφωνούν ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Θα δούμε. Φυσικά θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους συζητητές και με τη διαπραγματευτική ομάδα. Εγώ προσωπικά ε, συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε κάπως τη διαδικασία. Αλλά εννοείται το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει αρκετό χρόνο στην ε, διάθεσή τους να εξετάσουν και τους συμβιβασμούς και την τελική μας θέση. Αυτά για τις συστήσεις. Μήπως μπορέσουμε να κερδίσουμε κανένα μήνα δηλαδή. Αυτό εννοώ μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ό,τι νότερο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε γέρος. Καλώς. Περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα. Και πρώτον έχουμε το quick fix Μύθιτ. Είναι κάτι που τα συζητήσαμε βέβαια ήδη και χθε. Ε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο διαδικασία. Η συνεδρία των συντονιστών στο Στρασβούργο είχε συμφωνήσει μια διαδικασία για να προετοιμάσουμε τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις για να μπορεί εγκαίρωση κάθε πολιτική ομάδα να τις εξετάσει και να προετοιμάσει ένα κατάλογο ψηφοφορίας. Και όπως σας έγραψα χτες το βράδυ, με την πρώτη ευκαιρία παραβιάσαμε χτες ε, την προθεσμία και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εφαρμόσετε αυτούς τους κανόνες ε, με το να αναβάλλετε την ψηφοφορία για το δεύτερο θέμα που θα ψηφίσουμε, το φορολογικό. Πρέπει να τηρήσουμε τη διαδικασία γιατί οι ομάδες, ειδικά οι μικρότερες, δεν μπορούν να διαμορφώσουν ε, θέση όταν έρχονται τόσο αργά οι συμβαστικές προτάσεις. Οπότε δεν είναι επί της... Ε, είναι επί της διαδικασίας με το άρθρο 185, μάλιστα. Το ίδιο και η πράσινη και η γκουε. Μάλιστα και στην περίπτωση αναβολής είναι ένας υπέρ και κάποιος ομιλητής κατά. Λοιπόν, ε, να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπατε γιατί δεν είναι ακριβώς σωστό. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο συζητήσαμε την Πέμπτη δεν είναι διαδικασία, είναι μια κατευθυντήρια γραμμή και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα στην Επιτροπή μας ακριβώς γιατί εγκρίθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Και απαιτείται μια σταδιακή εισαγωγή για να προσαρμόσουμε αυτή την ψηφοφορία θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν οργανώσει τις ομάδες εργασίας ή ε, οι ε, την ίδια την ημέρα της συνεδρίασης στο Στρασβούργο. Αλλά αυτή είναι τυπική απάντηση βεβαίω ότι δεν ισχύει ακόμα. Η ουσία είναι ότι έχει μοιραστεί ο κατάλογος των ψηφοφοριών χτες 3 η ώρα το απόγευμα. Μετά έγινε μια συζήτηση και στην συζήτηση αυτή ζητήθηκαν κάποιες προσαρμογές και πολύ μικρές αλλαγές και με βάση τη συζήτηση στην Επιτροπή μας ο εισαγωγής, ε, εισηγητή, με συγχωρείτε, τι έκανε για να υπάρχει ευρύτερη πλειοψηφία όπω ζητήθηκε και προέκυψε από τη συζήτηση. Και είναι ελάχιστε οι αλλαγέ αυτέ. Ένα αριθμό, μία πρόταση και μία λέξη σε τρει συμβαστικέ προτάσει. Δεν επηρεάζει λοιπόν καθόλου την δομή των συμβαστικών προτάσεων και του καταλόγου ψηφοφοριών. Και μάλιστα και ο νέος κατάλογος ε, των ψηφοφοριών μοιράστηκε 6 ώρα το απόγευμα, εγκαίρος δηλαδή Θεωρώ λοιπόν πως εδώ πέρα σεβόμαστε την κατευθυντήρια γραμμή, η οποία όπως σας είπα ακόμα δεν ε, είναι ενισχύ. Οπότε νομίζω, βεβαίω εντάξει, είναι θεμητό μια πολιτική ομάδα να ζητάει αναβολή, αλλά δεν έχει κάποια νομική βάση, είναι πολιτικό αίτημα. Ε, το οποίο βεβαίω θα τεθεί σε ψηφοφορία. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε τώρα να τοποθετηθεί κατά αυτού του αιτήματο αναβολή. Υποθέτω, ναι, Ένα υπέρ πρώτα, ο κύριο Γκίγκολτ. Λοιπόν, Ρομπέρτο, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να πω πως ε, ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η συμφωνία μας, ότι είχαμε πει να μην υπάρχουν ε, μεγάλες αλλαγέ, να μην υπάρχουν αλλαγέ μετά τις 3 το απόγευμα τη προηγούμενη. Εσείς λέτε πως οι αλλαγέ αυτές ε, δεν έχουν σημασία. Για μας ε, κάνουν μεγάλη διαφορά στην ουσία, γιατί τώρα όσον αφορά την έκπτωση των τόκων έχουμε ασθενέστερη θέση από αυτή την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την συζήτηση της ΕΠΑ για το θέμα αυτό ακριβώς και τώρα δεν γνωρίζουμε πώς ε, θα θέλαμε να ψηφίσουμε. Θέλουμε να το συζητήσουμε εντός της ομάδας μας. Γι' αυτό ακριβώς συμφώνησαν οι συντονιστές για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό ζητά από τους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην ε, συνάντηση των συντονιστών να αναβληθεί η ψηφοφορία για να και να αποφεύγουμε τέτοιες αλλαγές τελευταία τελευταίας για ζητήματα ουσίας που είπαμε ότι δεν θα ξαναγίνονται. Δεν είναι νομικό το ζήτημα, είναι θέμα συνεργασίας. Και κύριε Πρόεδρε, ε, από εσάς θα περίμενα να υπερασπιστείτε αυτή τη συμφωνία και όχι να βρίσκετε επιχειρήματα ε, εναντίον. Και ειλικρινά απογοητεύομαι που παραβιάστηκε τόσο γρήγορα κανόνα. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο, δεν είναι η δικιά μου δουλειά να υπερασπίζομαι την ουσία ε, των πολιτικών συμβασμών παρά μόνο την διαδικασία. Και την ευκαιρία βεβαίω να ψηφίσει το Κοινοβούλιο μια θέση πριν το αυριανό ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί αν είναι να ακουστεί το Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πριν ε, τεθεί το θέμα στο ΕΚΟΦΗΝ, αλλιώς ε, προκαταλαμβάνουμε ολόκληρη την ε, διαδικασία. Λοιπόν, ποιος θέλει τώρα να τοποθετηθεί κατά της αναβολής. Ελίζα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες κάποιων ομάδων, αλλά πρέπει να έχουμε και κοινή λογική όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να κυρώσουμε όλη την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων που προηγείται της ψηφοφορία και δικαίως. Όλοι λοιπόν γνώριζαν το τι διακυβεύεται. Χθες έγινε η συζήτηση. Είτε λοιπόν παγων οι, θέση μας, θέσεις μας δύο-τρεις μέρες πριν ε, και δεν έχει νόημα να γίνει κάποια συζήτηση πριν από την ε, ψηφοφορία γιατί μετά οι θέσεις μας είναι άκαμπτες εντελώς ή αφήνουμε κάποιο περιθώριο ε, ελιγμών για συμβιβασμούς που μπορούν και πρέπει να συμβαίνουν μετά από τις συζητήσεις. Αυτό είναι το νόημα της συζήτησης. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και ο περιορισμός που αναφέρατε προσπαθούμε να επιταχύνουμε για κάποιο σκοπό συγκεκριμένο και νομίζω πως το πνεύμα ε, γίνεται σεβαστό. Δεν θεωρώ εγώ πως παραβιάζουμε κάποιον ε, κανόναν. Λοιπόν, μίλησε κάποιος υπέρ της αναβολής ε, και κατά. Μπορούμε τώρα λοιπόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Α, πρέπει να δοκιμάσουμε πρώτα το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία, ε. Δεν ψηφίζουμε. λοιπόν, τώρα Ψηφίζουμε το αίτημα αναβολής. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής. Όποιος θέλει να ψηφίσουμε τώρα ψηφίζει όχι. Όποιος θέλει αναβολή ψηφίζει ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, μη φιρ, πρώτα απ' όλα. Με βάση τις διαπραγματεύσεις, άρθρο 73.5. φιντ, πρώτα απ' όλα, Quick Fix. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική. Υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις. Πέρας. Δεκτή. Μη λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Όπως είπα και χθες ήταν επίτευγμα το ότι συμφωνήσαμε σε μια γρήγορη λύση σε τόσο περίπλοκα ζητήματα όπως το ΜΥΦΙΤ και το ΜΥΦΙΡ. Τώρα περνάμε. Να βρω τα χαρτιά μου. λοιπόν, έκθεση κανόνες κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν την, την ε, λειτουργία της ειδικής αγοράς. 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ, κατά, αποχές, να την επαληθεύσουμε, νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Να την απολυθεύσουμε. Ακόμα δεν έχει ψηφίσει κάποιος. Ωραία, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α με έτοιμα χωριστής ε, ψηφοφορίας σε έξι μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά έχει συγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος. Να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μέρος τέταρτο υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε και αυτό. Να έρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχουν ψηφίσει δύο συνάδελφοι. Εγκρίνεται. Μέρος πέμπτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το επαληθεύσουμε. Να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται μέρος. Έκτο υπέρ. χωριστή ψηφοφορία για την 116 που ζήτησαν οι πράσινοι. Ναι, έπρεπε να το έχω διευκρινίσει. Υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. έχει την ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. Περνάμε άρα στην τροπολογία 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική β με προφορική τροπολογία των πρασίνων πρώτο ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα σε δύο μέρη τη συμβαστική β. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 127. Την επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 132 υπέρ κατά πρέπει να είναι το ίδιο, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 142, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα με προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική γάμα χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε ωραία λοιπόν ψηφίζουμε τη συμβαστική γάμα αρχή τη ψηφοφορία Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί. Ωραία. Πέρας. Με ευρία πλειοψηφία. 148 υπέρ. Κατά αποχές. Α, συγγνώμη, δεν είδα το ΕΛΚ. 148 υπέρ. Ναι, να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά εποχές δεκτή. Συμβαστική ε. Πρώτα με προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. εποχές δεκτή. 153 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 154 υπέρ, κατά, 154, να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 155. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 157 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 158 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε την 158. Άρχεται η ψηφοφορία. Ακόμα δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 160 υπέρ κατά. Να επαληθεύσουμε την 160 αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μια ψηφοδιαφορά. 161 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε τα 161. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. 162 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, να την επαληθεύσουμε όμως. Ακόμα τέσσερις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Κατά οι σοσιαλδημοκράτες. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 166. ένας συνάδελφος ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Ε, συγκεντρωθείτε. 167 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Περίεργος συνδυασμός. Άρχεται η ψηφοφορία. 168. Έχετε συν. Εσείς στην 168. Μάλιστα. Εγώ βλέπω άλλο στο κατάλογο. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 171. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 175 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά να έλεγχος για το 21 πέρας και εγκρίνεται συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το 25 ψηφίζουμε πέρας Εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 186. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 189. Υπέρ. Οι άλλες πίπτουν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά ηλεκτρονικός σύνεχος για το 193 ψηφίζουμε πέρας και απορρίπτεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος το 194 ψηφίζουμε ακόμη ένας να ψηφίσει πέρασε εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 201. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ακόμη ένας συνάδελφος. Πέρασε. Και εγκρίνεται. 203. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 203. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική H. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 212. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά κάνουμε έλεγχο Άλλοι δύο. Πέρασε. Συμβαστική J. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216. Υπέρ. Κατά. Λίγο για το 216 ψηφίζουμε. Άλλος ένας. Πέρασε. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 218. Ψηφίζουμε. Άλλος ένας πέρασε. Και εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά. Νομίζω εγκρίνεται ας κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. εγκρινεται 223. υπέρ. Κατά. Δεν έχετε σηκώσει τα χέρια σας εύκρινος έλεγχος για το 2023. Πέρασε. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο, μια που δεν σηκώνετε τα χέρια σα, ε, να είναι σαφέ. Έλεγχο. Άλλο ένα πέρα. Ε, εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Ε, εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 236 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 236. Ψηφίζουμε. Άλλοι δύο. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται 52, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 53, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 54, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 54, ψηφίζουμε. Άλλοι δύο. Άλλοι δύο. Πέρασε. Α, απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική, 1. Χωριστή ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική όμικρον. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε για τη συμβαστική όμικρον δεύτερο τμήμα. Πέρασε. Εβδομήντα υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος για το εβδομήντα. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω για το ΕΛΚ. Καλώς πέρασε. Και εγκρίνεται 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Π. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 76. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω ψήφισε από το ΕΛΚ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική Κιού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. έλεγος για το 86. Ψηφίζουμε. Ας παραπάνω από το ΕΛΚ έχει ψηφίσει. Πέρασε. Εγκρίνεται. 87. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη. Αρ. σύγε τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε έλεγχο για το τρίτο τμήμα. Α, υπάρχει και τέταρτο τμήμα. Τώρα ψηφίζουμε για το τρίτο. Άλλοι δύο να ψηφίσουν. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, θα κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω από το έλεγχο Πέρασε. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές. Πάμε στη συμβαστική S, υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική T, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. V συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 ε, υπέρ κατά έλεγχος για το 99 ψηφίζουμε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 διότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την τοποθέτηση της πολιτικής μας ομάδας. Σας δίνω ένα πεντάλεπτο, λέει ο πρόεδρος. Έχετε πέντε λεπτά διάλειμμα, διακοπή. Grazie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

Ευχαριστώ.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 έτοιμοι. καλώ. Ψηφίζουμε για το τοπομένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία όμως. Ψηφίστε παρακαλώ. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω ψηφίζει. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Αλλά ίσως Ναι, έναν παραπάνω έχουμε. Έναν παραπάνω. Ένα από το ΕΛΚ δεν πρέπει να ψηφίζει. Ωραία. Τέλος τη ψηφοφορία. 18 συγγνώμη υπέρ, 14 κατά, 24 αποχέ. Τώρα νομοθετικό κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Πάλι έχουμε έναν από το ΕΛΚ παραπάνω. Πέρα τη ψηφοφορία. 20 υπέρ, 15 κατά, 21 αποχές. Εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κύριε Λάμπερτς, έχετε το λόγο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το επιχείρημά σας ότι πρέπει να καταψεφίσουμε για το κοφίν, δεν νομίζω ότι το κοφίν θα εντυπωσιαστεί από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν ήταν ε, καλή παρατήρηση κατά τη γνώμη μου. Η πλειοψηφία είναι η πλειοψηφία. Και έχουμε ένα κείμενο το οποίο υπερψηφίστηκε. Τελείωσε. Chairman. Mr. Luke? Yes. I would like just to announce that... Κύριος Λούκε. Ε, επικαλούμε το άρθρο 56 του κανονισμού για να εισαχθεί η ψήφος της μειοψηφίας η οποία αφορά την έκπτωση των τόκων ε, που θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε απαραίτητους επιχειρηματικούς σκοπούς. Επίσης κάποιες προτάσεις δεν εξετάστηκαν σωστά από την Επιτροπή αφού δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Σας ευχαριστώ, το σημειώνουμε. Ωραία. Λύεται η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση 30 του μηνός 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρίαση.